Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ετοιμαστείτε για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ετοιμάστε τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Αν μπορείτε να διακόψετε τις συζητήσεις μεταξύ σας, ιδίως οι επισκέπτες, So, ich bitte noch mal alle Kollegen, die Plätze einzunehmen und die Gespräche. Παρακαλώ, καθίστε, κάντε ησυχία και παρακαλώ να αποχωρήσουν οι μη έχοντες εργασία. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε. Αλλάξαμε χθε τη σειρά ψηφοφορία και θα ξεκινήσουμε με γάτες, σκύλους και νηφίτσες. Θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία για το σημείο 13. σκύλοι, γάτες και κουνάβια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υγειονομικές απαιτήσει. Αρχίζει η ψηφοφορία. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. είναι το σύντομο έγγραφο το, για το υπαριθμό 13. Εψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 33 υπέρ, 10 κατά. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. το σύντομο, το σύντομο έγγραφο. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν για γάτες, σκύλους και κουνάδια. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 49 υπέρ, καμία ψήφο κατά, καμία αποχή. Μάριο οποίο ζήτησε το λόγο. Έχω ξεχάσει την κάρτα μου. Αλλά φτάνει, καταφτάνει. Καλώ το σημειώσαμε. Και περνάμε στο σημείο 12, μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς. Ξεκινάμε με την τροπολογία 19. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 19. Εψήφισαν όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνεται. 20 έχει αποσυρθεί, 21 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπερίθμων 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε περνάμε γρήγορα στην τροπολογία 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 185 υπέρ, κατά, αποχές, Α, δεν είναι ξεκάθαρο να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Για την 185 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρυσι ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε για το 186, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 186. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 25 ψήφοι υπέρ, 30 ψήφοι κατά και μία αποχή. 187 ψήφοι υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 189. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 189 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 32 υπέρ, 26 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν η 189. Η 188 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44 υπέρ,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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 191 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 191 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 33 υπέρ, 28 κατά, εγκρίνεται. 59 υπέρ, 59 καταπίπτει, συγγνώμη, 59 καταπίπτει, ψηφίζουμε για την 60 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 με προφορική τροπολογία, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ,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 για την 193 με προφορική τροπολογία να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 38 κατά, απορρίπτεται. 72 και 194 απεσύρθησαν. Στην 196 έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεν είναι ξεκάθαρο ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 196 πρώτο τμήμα ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται εψήφισαν όλοι πέρασε τη ψηφοφορίας 27 υπέρ 33 κατά μία αποχή απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Α, καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Και περνάμε στην 195 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 195 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 31 ψήφοι υπέρ, 30 ψήφοι κατά. Συγχαρητήρια στους συντάκτες της γνωμοδότησης εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές. Μάλλον να ψηφίσουμε για την 74, επαναλαμβάνω, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 211 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για αυτή. Είναι 198 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 201, 202, 203 είναι ίδιες οι τροπολογίες. Μαζί ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Μόνο 10-15 συνάδελφοι συμμετέσχουν σε αυτή την ψηφοφορία. Στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Γιατί 201, 202 και 203 ηλεκτρονικός έλεγχος. Εψήφισαν όλοι. Πέραση τη προφορίας. Εγκρίνονται 32 ψήφοι υπέρ, 29 κατά. 199 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Για την 78 επαναλαμβάνω υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ κατά Αποχές. Μου λένε ότι μάλλον πρέπει να το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 204. Εψήφισαν όλοι. πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 24 υπέρ, 38 κατά. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 206. Να ελέγξουμε και τη 205. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για τη 205. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 26 κατά. Εγκρίνεται. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 207 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 210 υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 210. Εψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 34 κατά. Απορρίπτεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 83. Υπέρ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 73 δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. 90 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 212 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 101 δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. 95 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 213 καταβίπτει. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είμαι σίγουρος. Ελέγχουμε την 214 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Ένα παραπάνω από το ΕΛΚ. Πέρασε τη ψηφοφορία. 28 υπέρ, 34 κατά. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ, δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. 103 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 112 δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 215 υπέρ κατά 215 215 η 216 απερίφθη και ψηφίζουμε τη 215 τώρα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 κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 217, 218 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 219 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά... Να, ελέγξουμε τη 219 ηλεκτρονικά, έρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 29 κατά, εγκρίνεται. 128 υπέρ,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 κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 140. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορία. 139 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143. Και, και οι 220 είναι ίδιε. Ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 221 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εδώ ακούω θόρυβο. Κάποιος, ε, δεν ξέρω τι συζητάνε. συζητάνε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 221. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. 38 υπέρ 25 κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 145, περνάμε στην 146 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 του εισηγητού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ, κατά Αποχές απορρίπτεται. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 163 υπέρ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 Απεσύρθη 168 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία την 169. να ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Τώρα εντάξει. 37 υπέρ 27 κατά εγκρίνεται. 170, 171 είναι ίδιες, ψηφίζουμε μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 174 και οι 15 είναι ίδιες, μαζί ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές Καλύτερα να το ελέγξουμε. Τις δύο τροπολογίες 174 και 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορία. 55 υπέρ, 7 κατά. Ξεκάθαρο ήταν το αποτέλεσμα. Υπέρ. Φτάσαμε στην τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ, 177, συγγνώμη, υπέρ. Την 177 ψηφίζουμε. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 63 υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Ομόφωνα εγκρίνεται. Και περνάμε στην πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Πλήρης αρμονία στην αίθουσα. Συγχαρητήρια στον κύριο Σνέλχερντ. Καμία ψήφο κατά, καμία αποχή, ομόφωνη έγκριση. Συγχαρητήρια. so Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για το ψήφισμα για την COP18, διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στην Τόχα. Ελπίζω να προσφέρουμε και εμείς κάτι στη διεθνή συζήτηση για την αλλαγή του κλίματος για να αλλάξει κάτι στην στασιμότητα. Έχουμε κάποιους στόχους που θα θέλαμε να επιτύχουμε και τώρα το Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο ελπίζουμε να κινηθεί κάτι. Ε, ας περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία ξεκινώντας με την τροπολογία 16 με προφορική τροπολογία Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. να ψηφίσουμε για την 21 ηλεκτρονικά για να το ελέγξουμε. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 32 κατά. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 καταπίπτει και 23 καταπίπτει. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία την 26. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 31 κατά εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. 29 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Γιατί δεν βλέπω από εδώ σίγουρα τι ψηφίσατε. Για την 29 λοιπόν εψήφισαν όλοι. πέρα της ψηφοφορία. 24 υπέρ, 38 κατά και μία αποχή. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ με μια προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε και χωρίς την προφορική τροπολογία. Την 32. Να ελέγξουμε. Λοιπόν, ελέγχουμε την 32 με προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 32 εγκρίνεται με την προφορική τροπολογία. Δεν το είχαμε δει σωστά λοιπόν πριν. 31 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, Ελέγχουμε την 34 ηλεκτρονικά. 34. Εψήφισαν όλοι. πέρα της ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 28 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 Dan Jorgensen σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. να ελέγξουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 38. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 32 ψήφοι υπέρ, 31 ψήφοι κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 καταπίπτει, 40 καταπίπτει, 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 σε τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, Α, δεν μπορώ να δω σίγουρα. Να ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της 42 ηλεκτρονικά. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορία. 34 υπέρ 28 κατά μία αποχή. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε και το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά, γιατί δεν το βλέπουμε σωστά. Δεν το βλέπουμε, επομένως ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Για το δεύτερο τμήμα, 24 υπέρ, 38 κατά, απορρίπτεται. 43 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46, πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Για το δεύτερο τμήμα της 46, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι.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 Αποκλείεται, λέει ο Καλ Σουίτερ. Τώρα είμαστε εντάξει. 56 υπέρ, 7 κατά. Σαφώς εγκρίνεται. 51 υπέρ. Τη 49 θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά και τη 49. Ελέγχουμε τη 49 ηλεκτρονικά. Εψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. 30 υπέρ και 30 κατά. Απορρίπτεται. Ε, δεν μπορούμε να ψηφίζουμε μέχρι να περάσει. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο. 51 ηλεκτρονικός έλεγχος. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. «32 υπέρ, 29 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, να ελέγξουμε την 56. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 56. Εψήφισαν όλοι. πέρα στις πληροφορία. 32 υπέρ, 31 κατά. Εγκρίνεται. 59 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές για την 58 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία εψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας 34 υπέρ 30 κατά εγκρίνεται ΔΕΒΕ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΔΕΒΕ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 64 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Ψηφίζουμε για την 64 Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 30 υπέρ, 33 κατά μία αποχή. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα της 64. ΔΕΒΕ 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΔΕΒΕ 6 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, να ελέγξουμε την ΔΕΒΕ 6 δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορίες; 30 υπέρ, 34 κατα απορείτε. απορρίπτεται. ΔΒ1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΒ11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΒ10 υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγχουμε την ΔΒ10 ηλεκτρονικά. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 30 κατά εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 12 υπέρ, κατά, Αποχές. Ελέγχουμε την ΤΕΒΕ 12. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 33 υπέρ, 29 κατά και μία αποχή εγκρίνεται. ΤΕΒΕ 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ΤΕΒΕ 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ΤΕΒΕ 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε την αρχική τροπολογία χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 75 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα με ηλεκτρονική ψηφοφορία. 75 δεύτερο τμήμα. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 31 υπέρ 32 κατά. Με μικρή πλειοψηφία απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Οι φιλελεύθεροι δεν ψήφισαν. Δεν έχετε άποψη από αυτού. Το δεύτερο τμήμα της 78 το ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Εψήφισαν όλοι. Πέρας τη ψηφοφορία. 31 ψήφοι υπέρ, 32 κατά και μία αποχή απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 81 έχει ήδη εγκριθεί 84 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 84 δεύτερο τμήμα. Εψήφισαν όλοι. πέρα τη ψηφοφορία. 29 υπέρ, απορρίπτεται. 85, δύο τμήματα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 86 έχει ήδη εγκριθεί. Περνάμε στην 91 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 99 δύο τμήματα.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 106 ist auch 106 είχε επίσης εγκριθεί. ΔΕΒΕ 8 υπέρ, κατά, αποχές. Όχι, δεν είναι ξεκάθαρο για την ΔΕΒΕ 8, ηλεκτρονική επαλήθευση για την ΔΕΒΕ 8. Εψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 31 ψήφοι κατά, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 9 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 114 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εποχές Ε, δεν είναι ξεκάθαρο. 114 δεύτερο με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. πέρασε τη ψηφοφορία. 30 υπέρ, 34 κατά, απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 119 υπέρ. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 118. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 118. Δεν ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 120. Πάλι κατά τμήματα. Για το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 120. Εψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. 31 ψήφοι υπέρ, 33 κατά απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές. Να επαληθεύσουμε και την 121 ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι πέρασε τις ψηφοφορίες. 33 υπέρ, 31 κατά. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται επαλήθευση. Αν θέλετε να το επαληθεύσουμε. 122 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. 33 κατά. Απορρίπτεται. 29 υπέρ και μία αποχή. Ντεβε 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Ντεβε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ντεβε 3 Εγκρίνεται. Devastation 4. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά για το δεύτερο τμήμα της 2 ηλεκτρονική επαλήθευση. Εψήφισαν όλοι πέρα τις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ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 Εγκρίνεται ξεκάθαρα 55 ψήφοι υπέρ και 8 κατά. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεβε α υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε τη 15, ηλεκτρονικός έλεγχος. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορίας. 31 ψήφι. υπέρ, 32 κατά. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ Α υπέρ, κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την ΔΕΒΕ Α. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η ΔΕΒΕ Β τώρα υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεβε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεβε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεβε ε. υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. Επαληθεύουμε την ε, ΔΔΕ. Ε. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται η ΔΔΕ. ΔΔΕ ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την F. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 33 υπέρ, 29 κατά, εγκρίνεται. Δεβε G υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 54 υπέρ, 7 κατά, με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται αυτό το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Wir kommen zum Bericht von Anna Έκθεση της Άννα Ρόσπαχ τώρα. Θα ψηφίσουμε. Τροπολογία 32 πρώτα. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 1. 32. 32 τι είπατε, θέλετε ονομαστική, μάλλον θέλετε ηλεκτρονική, ναι. Πέρα τη ψηφοφορία. 37 υπέρ. 23 κατά. Εγκρίνεται. Άγκρι 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 κατά πίπτη, 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 31. Ψηφίστε παρακαλώ. Η 30 καταπίπτει είπαμε, γιατί εγκρίθηκε η άγκρη 1. «31. Θέλετε να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Α, όχι. Εντάξει. Συνεπώς. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 κατά καταπίπτει. 36 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τις ψηφοφορίες. 39 υπέρ. 37 υπέρ κατά αποχές 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να παληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την 38. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 28 υπέρ, 32 κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. 56 επαναλαμβάνω υπέρ κατά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 ηλεκτρονική ψηφοφορία για να ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορία. 34 υπέρ, 26 κατά, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την 66. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 30 υπέρ, 32 κατά, απορρίπτεται. Ναι, βιάστηκα. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και συμβαστική 7. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74 κατά πίπτη. 75 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 81 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα για το πρώτο τμήμα της 81. Ψηφίσατε όλοι πέρα της 28 υπέρ, 30 κατά, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Λοιπόν, δεύτερο τμήμα. Δεν θα ψηφιστεί. 82 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ωραία, επαληθεύουμε για την 86. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 32 κατά, απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88 υπέρ, με προφορική τροποποίηση. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 23 καταπίπτει. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 107 να επαληθεύσουμε για την 106. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την 107 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη φοφορίας. 30 υπέρ, 31 ψήφι κατά. Μία αποχή απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε για την 115. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 34 υπέρ, 28 κατά. Εγκρίνεται. Εντάξει, όλοι κάνουν λάθος. 116 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Α, οι 2 καταπίπτει. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 5. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. απορρίπτεται 6 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική αριθμός 1. Α, να επαληθεύσουμε για την τροπολογία 8. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά λοιπόν παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, με μια προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Άγκρι 11. Καταπίπτει. 24 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την 24 του Χόρστο Σνέλχαρτ. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Το ΕΛΚ ψηφίζει με έναν παραπάνω από όσους πρέπει. Πάντα μια ψήφος παραπάνω από το ΕΛΚ. Τώρα είναι εντάξει. 35 υπέρ, 26 κατά. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Θα επαληθεύσουμε για την 27. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 36 υπέρ, 25 κατά. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 10 δεν την ψηφίζουμε. Άγκρι 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 21 υπέρ, Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τη 19. Ωραία, ψηφίζουμε για τη 19. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πάλι το ΕΛΚ ε, ψηφίζει με μια ψήφο παραπάνω. Εντάξει τώρα, 35 υπέρ, 25 κατά εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία τώρα. Ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 62 ψήφοι υπέρ, καμία αποχή, μία ψήφος κατά. Λέει Πρόεδρος, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, την κυρία Ρόσμπαχ. The nurses. Και περνάμε τώρα στην γνωμοδοτηση Ξεκινάμε με την τροπολογία 78. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 83 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 29 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Όχι, 6 και 84. Είναι... Α, καταπίπτουν και οι δύο. 7. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ενοποιημένη τροπολογία 3 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89, 91, συγγνώμη, 91 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 12. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενωπημένη τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ Α, συγγνώμη, 100 όχι 10, 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ενωπημένη τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ενωπημένη τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ενωπημένη τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην 110 με μια προφορική τροπολογία. Μόνο με την προφορική τροπολογία δεν έχει δύο τμήματα. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο. Θα επαληθεύσουμε για την 24 ηλεκτρονικά. Εψήφισαν όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 39 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται με ξεκάθαρη πλειοψηφία. 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 114 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 35 υπέρ, 24 κατά μία αποχή. Ενοποιημένη τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 8 ηλεκτρονικά. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 48 υπέρ, 12 κατά, μία αποχή. Ξεκάθαρη πλειοψηφία εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε την 35 ηλεκτρονικά. Εψήφισαν όλοι πέρασε Εγκρίνεται η 35. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 123. Εψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται ξεκάθαρα η 123 και περνάμε στην 40 υπέρ. Κατά.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε λοιπόν την 50 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αψήφισαν όλοι. Απορρίπτεται. Να έχετε εμπιστοσύνη στον πρόεδρό σας. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά να το ελέγξουμε για την 126. Εψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 39 υπέρ, σαφώ εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ενωπημένη τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενωπημένη 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκαθαρό. Ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την 136. Εψήφισαν όλοι. Πέραση τη ψηφοφορία. 39 υπέρ 22 κατά. Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 140-141 είναι ίδιες, ψηφίζουμε μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε καλύτερα την 61 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, ψήφισαν όλοι, πέρας τις ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1 υπέρ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 2 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενοποιημένη 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 καταπίπτει και περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο. Τελική ψηφοφορία άρχεται λοιπόν. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 58 υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια στην Άνια Βάισκερβερ.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 Λοιπόν, ε, ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες, αγαπητοί συνάδελφοι, και σας ευχαριστώ πολύ για την προσεκτική σας συμμετοχή. Ολοκληρώσαμε αυτό το μαραθώνιο των ψηφοφοριών χάρη σε εσά. Και τώρα όσοι θέλουν να μείνουν για το σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης, να μείνουν παρακαλώ για να συζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γύρανση. Όσοι δεν θέλουν να μείνουν για το σημείο 15, παρακαλούνται να αποχωρήσουν συντόμως και ησύχως. Και ζητώ από την εισηγήτρια, η εισηγήτρια είναι η κυρία Λιωτάρ, και ζητώ από την εισηγήτρια να λάβει το λόγο μόλις υπάρξει λίγο ησυχία στην αίθουσα. Λιωτάρ. Η συγγήτρια, αν θέλει το λόγο βεβαίω, έχει το λόγο. Για το σημείο 15. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και συγγνώμη. Ε, δεν πρόσεχα για λίγο. Συζητούσαμε για την ψηφοφορία, βλέπετε, γι' αυτό.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 Χαίρομαι που είσαστε εδώ. Θα σας μιλήσω για μια έκθεση πρωτοβουλίας που ετοιμάζει η Επιτροπή μας και έχει να κάνει με την ανάπτυξη μιας, ε, ενός στρατηγικού σχεδίου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την ενεργό και την υγιή γύρανση. Βέβαια πολύ βαρύγδου πόσο όρος, περί τίνος όμως πρόκειται. Περί του εξής. Ο πληθυσμό στην Ευρώπη, και όχι μόνο, ζει περισσότερα χρόνια. Έχουμε δηλαδή μια γύρανση του πληθυσμού. Πράγμα το οποίο μας φέρνει μπροστά σε νέες προκλήσεις και πρέπει να προετοιμαστούμε και να προσαρμοστούμε σε αυτές. Σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει στην Επιτροπή μας αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας όπως σας είπα στην οποία αναφέρουμε διάφορα στοιχεία τα οποία μπορούμε και να συζητήσουμε στην Επιτροπή μας και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την γύραση του πληθυσμού με ποιο τρόπο δηλαδή γερνά και πώς ζει ο πληθυσμός αυτός. Βέβαια εδώ βλέπω αρκετού νέου στην αίθουσα. Μπορεί να νιώθετε ότι δεν σα αφορά το θέμα, αλλά να ξέρετε ότι όταν μιλάμε για την υγιή και την ενεργό γύρανση, αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους ηλικιωμένου, γιατί η γύρανση ξεκινάει ακόμα και πριν από τη γέννηση του ανθρώπου και επηρεάζεται από ένα σωρό παράγοντε, περιβαλλοντικούς παράγοντε, για παράδειγμα, και εμείς στην Επιτροπή μας φυσικά πρέπει να διαφερθούμε όλους ιδιαίτερω για αυτούς τους παράγοντε, αλλά έχει να κάνει και με κοινωνικού και οικονομικού παράγοντε έχει να κάνει με την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στην κοινωνία, με την ασφάλεια των τροφίμων, με την αηφόρο ανάπτυξη. Έχει να κάνει βέβαια και με την πρόληψη στον τομέα της υγείας και με την εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας του πληθυσμού. Υποστηρίζω λοιπόν πάρα πολύ τον στόχο της Επιτροπής ε, προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν περισσότερα χρόνια κάτω από καλέ συνθήκες και είναι ένας στόχο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2020. Πιστεύω ότι είναι πολύ σωστό. Όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι θέλουμε να πετύχουμε ως στόχο υγείας. Η κοινωνία πρέπει να εμπλέκεται σε αυτόν τον στόχο για υγιή γύρανση. Δεν πρέπει δηλαδή να δούμε πολύ περιορισμένα το θέμα, αλλά να το δούμε ευρέως, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι οι ίδιοι που πρέπει να ασχοληθούν με αυτό, αλλά η κοινωνία ολόκληρη. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να μην τα συζητάμε μεταξύ μας τα θέματα αυτά που αφορούν τους ηλικιωμένους, αλλά να τα συζητάμε με τους ηλικιωμένους, για να δούμε αυτοί τι εννοούν όταν μιλούν για υγιή και ενεργό ε, γύρανση. Είναι πολύ καλό να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο για μένα βασίζεται σε τρει πυλώνες. Ο πρώτο πυλώνας έχει να κάνει με την πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την πρώιμη διάγνωση. Ο δεύτερο πυλώνας έχει να κάνει με την περίθαλψη και τη θεραπεία και ο τρίτο έχει να κάνει με την αναργό γύρανση και την ανεξάρτητη διαβίωση και τη συμμετοχή στην κοινωνία των ε, ηλικιωμένων. Όσον αφορά την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, θέλω να σας πω ότι όταν μιλάμε για την πρόληψη, εγώ έχω πάει σε πολλά συνέδρια και όταν ρωτάτε τι ξοδεύει κανείς για την πρόληψη στην υγεία, διαπιστώνεται ότι είναι το 3% του συνόλου. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό που πηγαίνει στην πρόληψη. Θα έπρεπε να επενδύουμε περισσότερο στην πρόληψη και όχι μόνο την πρόληψη ασθενειών, αλλά και την ε, βελτίωση του περιβάλλοντος, των σπιτιών μέσα στο οποίο ζούμε, των μεταφορών με τις οποίες μετακινούμαστε κτλ. Επιπλέον φαίνεται ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο κοινωνικό και οικονομικό στάτους των ανθρώπων και ε, την ε, ηλικία μέχρι την οποία φτάνουν. Δηλαδή πρέπει να επενδύουμε όχι μόνο στην περίθαλψη, αλλά να επενδύουμε και στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν οι άνθρωποι για να μπορούν περισσότερα χρόνια να ζουν καλά οι άνθρωποι αυτοί. Επιπλέον θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και τις διαφορές που υπάρχουν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Άλλες ε, περιφέρειες μπορούν να δουλέψουν καλύτερα στις μεταφορές, άλλες ε, ε, στον εθελοντισμό υπέρ των ηλικιωμένων και αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας στην δικιά μας την έκθεση. Και όσον αφορά την ε, ε, περίθαλψη επίσης να φροντίσουμε στο επίκεντρο αυτής να βρίσκεται ο άνθρωπος, ο πελάτης ασθενής κατά κάποιο τρόπο. Οι ηλικιωμένοι λέμε συχνά ότι κοστίζουν πάρα πολλά στην κοινωνία. Δεν είναι όμως πάντοτε ε, οι ηλικιωμένοι που αναλαμβάνουν το κόστος πρέπει να είναι η κοινωνία, ολόκληρη η κοινωνία. Θα έλεγα μάλιστα ότι υπάρχει ο κίνδυνος ε, μερικές ε, φορές να μην έχουν αρκετούς οικονομικούς πόρους οι άνθρωποι και δεν συμβαίνει αυτό μόνο στις υποανάπτυκτες χώρες. Οι ηλικιωμένοι δεν τρέφονται καλά. Όχι μόνο λόγω των οικονομικών πόρων που τους λείπουν όπως σας είπα, αλλά γιατί ε, μερικές φορές ε, χάνουν τη γεύση τους ή δεν τους αρέσουν αυτά που τρώνε οι άλλοι μέσα στην οικογένειά τους, αν ζουν στην οικογένειά τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, τους οποίους εμείς πρέπει να μελετήσουμε. Γιατί όσο δεν τους μελετούμε και δεν διορθώνουμε την κατάσταση, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δεν τρέφονται, οι ηλικιωμένοι, καταλήγουν στα νοσοκομεία, κάτι το οποίο κοστίζει πολλά λεφτά στην κοινωνία. Το τελευταίο το οποίο αναφέρομαι στην έκθεσή μου είναι η ανεξάρτητη διαβίωση. Πάρα πολλοί ηλικιωμένοι έχουν πει ότι θέλουν όσο γίνεται περισσότερο να ζουν ανεξάρτητοι μόνοι τους ε, στο σπίτι τους. Άρα το περιβάλλον πρέπει να προσαρμοστεί στην ανάγκη αυτή. Το να ζει κάποιος ανεξάρτητος δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζει και απομονωμένος. Είναι πολύ βασικό αυτό για την κοινωνία. Η κοινωνία δηλαδή πρέπει να προβεί στις αλλαγές που χρειάζεται έτσι ώστε οι ηλικιωμένοι να μπορούν να διαβιώνουν ανεξάρτητα χωρίς όμως να είναι απομονωμένοι. Φυσικά έχω γράψει πάρα πολλά πράγματα στην έκθεσή μου, μπορείτε να τα διαβάσετε με την ησυχία σας, αλλά είμαι πάρα πολύ περίεργη πραγματικά να μου πείτε τι γνώμη έχετε, τι παρατηρήσεις έχετε και τι σχόλια έχετε να κάνετε στο όσο έχω γράψει μέχρι τώρα. Να ξέρετε ότι θα τα λάβω υπόψη μου, θα μελετήσω τις προτάσεις σας και θα έρθω με νέες δικές μου προτάσεις στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στην σκιώδη εισηγήτρια από το ΕΛΚ, στην συνάδελφο Αντωνέσκου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια για την έκθεσή της και την παρουσίασή της. Νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε πολύ περισσότερο το θέμα της ε, διάγνωσης. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το, να δούμε το θέμα του υγιεινού τρόπου ζωής. Αυτό θα βοηθήσει πολύ σε υγιή και ενεργό διαβίωση και γύρανση. Διότι πολλές ασθένειες εξελίσσονται πολύ αργά και όταν φτάσει κανείς στην τρίτη ηλικία είναι πολύ αργά να κάνει κάτι. Οφείλονται στον τρόπο ζωής τα προηγούμενα χρόνια. Άρα πρέπει να δούμε την γύρανση σαν μια διαδικασία πράγματι που διαρκεί ολόκληρη τη ζωή. Είναι επίσης σημαντικό να δούμε και τι έρευνα γίνεται και στον φαρμακευτικό τομέα, στη θεραπεία δηλαδή. Να λάβουμε υπόψη μας πολλές διαστάσεις και την οικονομική και την κοινωνική διάσταση χρόνιων ασθενειών. Άρα η προσέγγιση μας πρέπει να είναι πολυδιάστατη. Να δούμε τι γίνεται στην έρευνα, στον τομέα της υγείας, γιατί Αν δεν ε, τα συνδέσετε όλα αυτά με το τι κάνει η κοινωνία και αν ε, δεν χρησιμοποιήσετε τις έρευνες που γίνονται σε άλλους τομείς και εδώ, τότε υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είναι πολυδιάστατη και πολυτομιακή η προσέγγισή μας και να χρησιμοποιήσουμε την έρευνα που έχει γίνει σε διάφορους τομείς και να τη χρησιμοποιήσουμε εδώ, στην υγεία στην φροντίδα και την περίθαλψη. Έπειτα πράγματι υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στις περιφέρειες, στις περιοχές, όσον αφορά την αντιμετώπιση των ηλικιωμένων και την υγεία. Για το δεύτερο πυλώνα, που είναι η περίθαλψη και η θεραπεία, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε επαρκές επίπεδο περίθαλψης και φροντίδας όταν ε, συμμετέχει η οικογένεια πρέπει να την στηρίζουμε. Ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε περισσότερο στην έκθεση για κέντρα περίθαλψης. Κάτι άλλο που με απασχολεί εδώ είναι το σημείο στο οποίο αναφέρεστε στην ανεργό γύρανση και την ανεξάρτητη διαβίωση. Πώς δηλαδή θα στηρίξουμε τα άτομα αυτά που θέλουν να ζουν ανεξάρτητα. Να λάβουμε υπόψη μας ότι πρόκειται και για ένα όφελος προς την κοινωνία όταν τα άτομα αυτά μπορούν πράγματι να ζήσουν ανεξάρτητα και όχι όμως απομονωμένα. Είναι κέρδος για όλους. Γι' αυτό και πρέπει να προωθήσουμε την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων. Να ζουν αυτοί οι άνθρωποι νιώθοντα ότι ανήκουν στην κοινωνία, ότι είναι και αυτοί οι μέλη της κοινωνίας. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν φτιάχνουμε μηχανισμούς για να πετύχουμε τους στόχους μας, που είναι η υγιή γύρανση. Από στρατηγική άποψη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι πρέπει να λάβει υπόψη τη περισσότερο τη συνέργεια μεταξύ διαφόρων πολιτικών και να βρει τρόπους να χρηματοδοτήσει τις προσπάθειές μας. Αυτές ήταν κάποιες σκέψεις που είχα. Και από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι θα υποβάλω και κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στον Μάριο Πυρίλο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Λιωτάρ για την εξαίρετη έκθεσή της. Το χρόνο αυτός που φτάνει στο τέλος του είναι ευρωπαϊκό έτος ε, δραστηριε Γύρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η έκθεση πρωτοβουλία συναδέλφου θα πρέπει λοιπόν να θέσει κάποια στιγμή την σύνδεση με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, αλλά και για να εκθέσει τις μελλοντικές προκλήσεις που αναμένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συγχαρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολήθηκε με το θέμα της δραστήριας γύρασης μαζί με την αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενναίες. Η αύξηση των ηλικιωμένων ανθρώπων στις περισσότερες φορές θεωρείται ως βάρος ε, που επιβαρύνει τους νεότερους και τους εργαζόμενους. Χάρη στις πρόοδους της ιατρικής σήμερα, Κανείς ζει πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν και, γι αυτό είναι σημαντικό, και σε καλύτερη κατάσταση και γι' αυτό είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να παραμείνει κανείς στη θέση απασχόλησης του. Ότι ηλικιωμένα άτομα είναι πολύτιμα. Η εμπειρία τους και η δεξιότητά τους που έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των ετών πρέπει να διαβαστεί στους νέους. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προωθήσει στοχευμένες δράσεις ώστε να υπάρξει μια επαφή ανάμεσα στις γενναίες τόσο για την απασχόληση των νέων και τη βοήθεια μέσω της βοήθειας προς τους ηλικιωμένους όσο και προς τις ε, ηλικιωμένους με μια πολιτική που θα ε, γνωστοποιήσει σε όλους ότι η δραστήρια γύρανση αφορά όλες τις γυναίες. Έτσι θα, πρέπει να σκεφτούμε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία μας. Παρεμβάσεις σε επίπεδο δημόσιων πολιτικών θα πρέπει να αναγνωρίζουν στην μακροβιότητα μια ευκαιρία και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις ε, πριν, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν και οι κοινωνικές προκλήσεις τη σήμερα. Θα ε, έχει τεθεί ο στόχος της αύξησης ε, κατά δύο έτη του αριθμού ετών σε καλή υγεία. Ε, με καλή υγεία. Ήδη αυτός ο φιλόδοξος στόχο, χρειάζεται ε, πόρους για να επιτευχθεί. Η σημερινή σοβούσα κρίση όμως έχει φέρει την δημόσια δίκηση σε πολλέ πολλές περικοπές, ε, ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Θα χρειαστεί μια διαδικασία βελτιστοποίησης των οικονομικών πόρων έτσι ώστε να παρέμβουμε για να εγγυηθούμε την σωματική, κοινωνική και ψυχολογική υγεία και που επιτρέπει στους ηλικιωμένους να παίξουν δραστήριο ρόλο και να έχουν μια ζωή ποιοτική και ανεξάρτητη. Να προωθήσουμε λοιπόν την δραστήρια γύρεση σημαίνει να δημιουργήσουμε καλύτερες ευκαιρίες έτσι ώστε γυναίκες και άνδρες ηλικιωμένοι να μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν ρόλο στην αγορά εργασίας, να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και τον κοινωνικό απολυτισμό, να ενθαρρύνουμε την εθελοντική, τον εθελοντισμό, τη συμμετοχή στην καθημερινή ζωή, καθώς και να προωθήσουμε την υγιή και αξιοπρεπή γύραση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Μάριο Πυρίλο και θα δώσω το λόγο για το ECR στην Julie Gerling. Um, ευχαριστώ. Εγώ μιλώ εξ ονόματος της Αν ε, Ρόσμπαχ που είναι η σκιώδης εισηγητριά μας και ε, μπορώ να συμφωνήσω με αρκετά από αυτά που υπόθηκαν. Είμαστε πεπισμένοι ότι χρειάζονται συνολικές μεταρρυθμίσεις ώστε να παρεμποδιστούν ε, σοβαρές ελλείψεις της αγοράς εργασίας αλλά να αναγνωρίσουμε επίσης ότι είναι πολύ κρίσιμες οι διαφορές, σε μεγάλες οι διαφορές. Ένα πρόσφατο ευρωβαρόμετρο ρώτησε τις κυβερνήσεις ε, κατά πόσο θα καθιστούσαν ε, πιο εύκολη την απασχόληση των γυρεών των ηλικιωμένων. Ε, πολλές διαφορές υπήρξαν στην Ολλανδία και στη Βρετανία έλεγε, έλεγαν ότι θα πρέπει να δουλεύουν περισσότερο οι γεροντότεροι ενώ στις νοτιότερε χώρες αυτό δεν ήταν, θεωρείται προτεραιότητα. Ε, θα έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις αν θέλουμε να φτιάξουμε ευρωπαϊκή πολιτική για το θέμα αυτό. Επίσης είδαμε ότι η ε, επίσημη ηλικία συνταξιδότηση προτείνεται να αναθεωρηθεί σε 24 από τις 34 ε, χώρες μέλη ε, δηλαδή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, προς τα πάνω κιόλας. Άρα έχουμε ένα σαφή στόχο, αλλά διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ε, θα πρέπει να τον επιτύχουμε σύμφωνα με την κοινωνία. Ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια μεταρρύθμιση του συστήματος συνταξιδότησης ώστε να είναι πιο καλά χρηματοδοτούμενο και ξέρουμε επίσης από την ίδια έκθεση του ΩΣΑ ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σκοπεύουν να αυξήσουν τις, τις κυβερνητικές για τις συντάξεις, σε ορισμένε περιπτώσεις και μέχρι και 15%. Τεράστια αλλαγή δηλαδή. Στηρίζουμε την συγγήτρια για το θέμα του, αύξηση, του στόχου αύξησης της υγιούς ζωής για δύο χρόνια, αλλά και πάλι είναι δημογραφική η πρόκληση αυτή, ανάλογα με το κράτος μόνος για το οποίο μιλάμε. Μια ερώτηση τώρα για την εισηγήτρια, αν μου επιτρέπετε. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε πώς θέλει να αντιμετωπίσει τα διαρθωτικά θέματα και πώς θα εξαλείψει τις ανισότητες λόγω ηλικίας. Θέλουμε να δούμε, είναι περίπλοκα τα θέματα, θέλουμε να δούμε τις τροπολογίες. Ρέστε Ρώση. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγχωρείτε, κανένα λάθος. Η Φρίντα Μπρέπολς πρώτα. Περίμενα σε εδώ από εδώ, Φρίντα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για τους πράσινους. Και εμείς ε, λοιπόν θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ευρεία συνένεση για το γεγονός ότι η δημογραφική γύρανση, η γύρανση του πληθυσμού μας δηλαδή, βάζει την κοινωνία μας μπροστά σε νέες προκλήσεις. Σωστά λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τις προτάσεις της που λένε ότι πρέπει να προσέξουμε και το κόστος το οποίο βαρινόμαστε εξαιτία αυτής της γύρανσης αλλά συγχρόνως έχουμε και την ευκαιρία να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων στις κοινωνίες μας έτσι ώστε να μπορούν ε, να γερνάνε με υγεία και με δραστηριότητες. Χρειάζεται λοιπόν ε, κάποια καινοτομία στον ε, τομέα της φροντίδας και της περίθαλψης. Και εδώ είναι που η ευρωπαϊκή αυτή σύμπραξη καινοτομία μπορεί να προσφέρει πολλά. Στην Φλάνδρα, για παράδειγμα, από που έρχομαι, έχουμε το Flanders Care, που είναι ένα πρόγραμμα με καινοτόμες προτάσεις για υπηρεσίες φροντίδας ποιότητας. Κάτι το οποίο βέβαια δίνει και κίνητρα στην οικονομία. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας να υπάρχει και η προοπτική της καινοτομίας στην ε, φροντίδα και την ε, περίθαλψη λαμβάνοντας υπόψη μας βέβαια το στόχο του 2020. Και όταν λέω καινοτομία, όχι μόνο για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της γύρανσης, αλλά με την καινοτομία μπορούμε να έχουμε γενικότερα ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Με την έκθεση αυτή πρωτοβουλίας φυσικά δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ενεργογύρανση. Όχι, πρέπει να επικεντρωθούμε στα πιο σημαντικά και να δούμε τι μπορεί να εφαρμοστεί και τι συγκεκριμένα αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Μ' άρεσε που διάβασα ότι η συγγήτρια συμφωνεί με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, σημασία έχει να επικεντρωθούμε στη σχέση που έχει η καινοτομία με την φροντίδα και η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη αυτή καινοτομία να ασχοληθεί ακριβώς με αυτό το θέμα. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να κάνω και κάποιες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπήρξε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 27 Ιουνίου και εκεί έλεγε μιλούσε για τη συμμετοχή των ε, εμπλεκόμενων. 361 σχέδια υπήρχαν. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί θα συμμετέχουν στην διάσκεψη που σήμερα λαμβάνει η χώρα. Θέλω να ξέρω λοιπόν πώς έχει προχωρήσει αυτό το θέμα. Δηλαδή, πώς θα πάρει ακριβώς μορφή αυτή η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας, πώς θα μπορέσουμε να, στην πράξη να καταλάβουμε τα αποτελέσματα. Έπειτα γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον έχει σκεφτεί καθόλου πώς θα γίνει αυτή η σύνδεση της καινοτομίας με την περίθαλψη. Έπειτα αυτή η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας πώς θα ενσωματωθεί σε όλες τις χώρες μέλη. Κατά τα άλλα, να ξέρετε ότι είμαστε διατεθειμένοι επικοδομητικά να συνεργαστούμε με την εισηγήτρια και τους άλλους κοιόδης εισηγητές. Τώρα, κύριος Ρώση. Ευχαριστώ. Ε, Πρόεδρε, είμαι πολύ ευνοϊκά διακείμενο στο κείμενο αυτής της έκθεσης και θα πρέπει να σας πω πως συμφωνώ με την εισηγήτρια. Απλά θα ήθελα να τη ρωτήσω αν υπάρχει τρόπος να προσθέσουμε ίσως με κάποια τροπολογία στις ε, αιτιολογήσεις το θέμα που σχετίζεται με την γύρανση που θα πρέπει να πω ότι στην Ευρώπη ευτυχώς, γιατί το βλέπουμε περισσότερο ευτυχώς, γιατί υπάρχουν λίγες γεννήσεις με χαμηλή γενετικότητα οδηγεί στην αύξηση των ε, ηλικιωμένων. Εγώ θα έλεγα πως ήταν καλύτερο να υπάρχουν και ε, υπηρεσίες προς την οικογένεια, γιατί πολύ συχνά ε, οι οικογένειες δεν κάνουν παιδιά γιατί δεν, μπορούν, δεν έχουν αρκετή στήριξη, αρκετή βοήθεια ε, τη στιγμή που η γυναίκα είναι ε, έγκυος ή σε άδεια μητρότητας. Οι υπηρεσίες λοιπόν για την οικογένεια είναι μια εξαίρετη λύση για να βελτιώσουμε το έλλειμμα το δημογραφικό της γυριάς μας Ευρώπης. Ε, τώρα, για τα υπόλοιπα προφανώς ε, μιλάμε για ηλεκτρονική υγεία και με καλύτερη υγεία και τα λοιπά, λίγα δαπανώνται και πρέπει να δαπανεθούν περισσότερο και ακόμα και αν πούμε ότι η πρόορη σύνταξη μάλλον η πρόορη, η έγκαιρη μάλλον διάγνωση, σημαίνει δαπάνη χωρίς να έχει ανακαλύψει μια ασθένεια. Αλλά αν την ανακαλύψω και την ανακαλύψω και την εντοπίσω και εγκαίρως, πέρα από την λύση και μπορώ, της, του προβλήματος και τη θεραπεία, μπορώ να έχω αποτελέσματα γρηγορότερα και με χαμηλότερο κόστος. Σκεφτούμε τι, πόσο κοστίζει μια παθολογία καρκίνου που έχει προχωρήσει για χρόνια και πόσο λιγότερο θα κόστιζε ακόμα και όσον αφορά την ποιότητα ζωής του ανθρώπου τρόπο αν ε, την έχει εντοπιστεί εγκαίρως ε, ή με μια διάγνωση ακόμα πιο προηγμένη ε, ας πούμε με το παράδειγμα που σας δίνω για το DNA να καταλάβουμε αμέσως ότι ένα παιδί ως, μεγά, ως ενήλικας μπορεί να έχει ε, να, υποφέρει από διάφορες ασθένειες και άρα να προλάβουμε με πολύ χαμηλότερο κόστος τις ασθένειες αυτές. Τώρα, βοήθεια και θεραπείες, οι αγωγές και εδώ ξεχνάμε και θα πρέπει να το βάλουμε εδώ ότι το πρόβλημα πολλών ηλικιωμένων είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουν και οι ε, τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Το να καταστούν οι πόλεις λοιπόν προσβάσιμες στα άτομα με ειδικέ ανάγκες ε, σημαίνει και να, ότι θα είναι και προσβάσιμες ε, για τους ηλικιωμένου, που συχνά έχουν λιγότερες ευκαιβολίες από ό,τι άλλοι γιατί έχουν κινητικές δυσκολίες, ε, προβλήματα για να πάνε στο θέατρο, να, πάνε, να βγουν στο εστιατόριο, να βγουν στο δρόμο γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουν το πι ή, μπαστονα, ή να μπαστούνι ή ακόμα και την αναπηρική καρέκλα. Πρέπει λοιπόν ε, οι πόλεις να σέβονται τα δικαιώματα των ε, ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες αλλά και όλων όσων ε, γερνούν. Να δοθούν λοιπόν υπηρεσίες που στις πόλεις βέβαια, αλλά και στα μικρά κέντρα, τους μικρούς κόμους, γιατί αν, αν και το έλεγε και η συγκέντρια, όλο και περισσότερο μετακινούμαστε προς τις πόλεις, που εκτός που εγκαταλείπουμε την Ήπεθρο, πολύ συχνά η ποιότητα ζωής μας είναι χειρότερη. Πολλέ φορές ζει κανεί σε ένα μικρό ε, αστικό κέντρο και από άποψη ποιότητα ζωή και από σωματική άποψη. Και ε, αν δώσουμε λοιπόν υπηρεσίε στα μικρά κέντρα, καλούμε τον ηλικιωμένο να μείνει στο σπίτι του όσο γίνεται πιο πολύ και να ζήσει και καλύτερα. Κλείνω με το αίτημα τη ε, εισηγήτρια, ώστε ενδεχομένω να αξιολογήσουμε κάποιε επιπλέον τροπολογίε σε αυτό το κείμενο και σα ευχαριστώ για τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Vielen Dank. Damit haben wir die σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο των σχεδόν ομιλητών. Υπάρχουν αρκετοί ομιλητέ που θα ήθελαν το λόγο. Θα σα διαβάσω το κατάλογο των ε, συναδέλφων που έχουν ζητήσει το λόγο. Dann Μήπω ξέχασα κανέναν? Όχι. Κλείνει λοιπόν ο κατάλογο των αγορητών και σας παρακαλώ μην ξεπεράσετε το 1,5 λεπτό, γιατί έχουμε άλλο ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη που πρέπει να ολοκληρώσουμε. Η κυρία Γκροστέτ. Πρόεδρε, για το πρώτο θέμα. Μία παρατήρηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εκπροσωπείται σε αυτή την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Κοινοτομίας για Ενεργό και Υγιή Γύρανση είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες, ο ιδιωτικό τομέα, οι επαγγελματίε υγεία, οι ε, κοινωνικοί εργαζόμενοι, οι εκπρόσωποι των ε, ηλικιωμένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμω όχι. Και αυτό είναι σφάλμα. Τώρα έρχομαι στην έκθεση αυτή καθεαυτή τη κυρία Λιωτάρ. Εγώ θα ήθελα να μιλάμε περισσότερο για την κοινοτομία, γιατί πρόκειται για μια ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομία για την ενεργό και υγιή γύρανση. Μια σύμπραξη λοιπόν όπου ζητάει προτάσεις για καινοτομία. Αυτό που διακυδεύεται εδώ είναι ακριβώς πιο ευφυής χρήση της καινοτομίας για να αντιμετωπιστεί πρόκληση της γύρανσης. Άρα θέλουμε προγράμματα καινοτομίας και στον τομέα της ε, κατάρτισης και της πληροφόρησης αλλά και των εργαλείων. Είτε πρόκειται για συστήματα πληροφορικής διαδραστικά προκειμένου να συνεχίζουν να ζουν στα σπίτια τους ηλικιωμένοι. Έπειτα όσον αφορά την περίθαλψη και τη θεραπεία πρέπει να ενισχύσουμε την έρευνα. Πολλές κλινικές δοκιμές έχουν γίνει ήδη αλλά δεν μας επέτρεψαν να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε ασθένειε που σχετίζονται με την γύρανση. Άρα η φαρμακευτική βιομηχανία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να συνεχίσει τι ερευνητικέ προσπάθειε. Γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε τη σχέση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για να στηρίξουμε την καινοτομία και να καταπολεμήσουμε τι ε, μάστιγε αυτέ που συνδέονται άμεσα με την γύρανση. Στηρίζω λοιπόν την πρόταση τη κυρία Λεωτάρα, αλλά θα υποβάλω κάποιε τροπολογίε για τα θέματα τα οποία μόλι έθιξα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γενικά προσπαθήσαμε Προσπαθήσαμε σε αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου να στείλουμε κάποιον εκπρόσωπο ε, κατόπιν αποφάσεως του Προεδρείου. θέλουμε να είναι εγγυημένη η ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου και θα θέλαμε να μην ε, γίνονται συζητήσεις πουθενά αλλού παρά μόνο εδώ. Εδώ να λαμβάνονται οι νομοθετικές αποφάσεις και γι' αυτό ε, απερίφθη αυτό το αίτημα. Συνάδελφος Γκουτιέρεθ. Ε, oh, ναι. Η κυρία Συμφωνώ με το ότι πρέπει να ξαναδούμε αυτό το θέμα. Γιατί να μην είμαστε στη steering ε, committee, στις επιτροπές αυτές ε, steering. Εγώ στηρίζω βέβαια την κυρία Λιωτάρ, την θέση της δηλαδή, αλλά υπάρχει κάτι που με απασχολεί. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα με ένα έγγραφο. Και το πρόβλημα της γύρανσης είναι περίπλοκο και τεράστιο. Γι' αυτό θα έπρεπε να προτείνουμε ένα πρόγραμμα, ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο να μπορούμε να παρακολουθούμε. Όπως ε, για το περιβάλλον, για την Ατζέντα ε, 2020. Να δούμε δηλαδή μέσα σε αυτό το πρόγραμμα τι κάνουν οι διάφορες χώρες και τι προτεραιότητες έχουν. Να υπάρχει ένα πρόγραμμα δηλαδή παρακολούθησης που θα θέσει τις προτεραιότητες μας για τα ηλικιωμένα άτομα. Άλλες χώρες έχουν τέτοια πράγματα, άλλες δεν έχουν. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Για παράδειγμα, η απομόνωση των ηλικιωμένων που δημιουργεί από μόνη τη τεράστια προβλήματα. Και υπάρχουν μελέτε που έχουν δείξει πόσο αρνητική επίπτωση έχει απομόνωση στην γύρανση του πληθυσμού, στην ποιότητα δηλαδή της γύρανσης, η κακή διατροφή των ηλικιωμένων. Έπειτα υπάρχουν τα μεγάλα τεχνολογικά λόμπι. Σήμερα, στην πρώτη σελίδα της International Herald Tribune λέει ότι μειώνεται το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξαιτία των λόμπι. Η τεχνολογική ουτοπία προσπαθεί να μας πείσει ότι θα λύσουμε τα προβλήματα των ηλικιωμένων μόνο με μηχανήματα. Προσοχή λοιπόν, έχουμε ως ορίζοντα το 2020 θέλουμε την καινοτομία να τη χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την ζωή των ηλικιωμένων. Αλλά υπάρχει και η τεχνολογική ουτοπία. Εγώ θα προτιμούσα οι συνάδελφοι να μιλάνε για την κοινωνική διάσταση περισσότερο. Η κυρία Χίμνερ, ένα μισή λεπτό παρακαλώ και εσείς όπως και οι προλαλήσαντες. Ε, ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. η κοινωνία μας γυράσκει και έχουμε όλοι αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Έχουμε μέλη της οικογένειάς μας που ε, γερνούν και εμείς οι ίδιοι γερνάμε. Είναι ένα κομμάτι της ζωής. Ε, η καλή ζωή είναι αυτή που βοηθά στην ε, υγιή και καλή γύρανση επίσης. Ε, θα πρέπει αυτό να το έχουμε ε, υπόψη μας. Δεν έχουμε αρκετούς επαγγελματίε δε για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, αλλά ούτε και για τη στήριξη των οικογενειών. Θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική αστικοποίηση. Και να εξετάσουμε τις δημογραφικές αυτές αλλαγές, να σκεφτούμε και αυτό το πρόβλημα. Η δραστήρια γύρανση. Αυτό είναι δυνατόν όταν έχουμε διαβίου μάθηση Κάποιες φορές ε, αυτές τις δραστηριότητες όπως ε, το Πανεπιστήμιο της Τρίτης ηλικία ε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ώστε να μπορέσει ο κόσμος να βγει και να κάνει κάτι στη ζωή του. Να γίνει η αναθεώρηση διαφόρων λύσεων στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό σύστημα. Η κυρία Κλάσια, ένα μισή λεπτό. Και εγώ όπως και οι άλλοι συνάδελφοι. Ξέρετε, καμιά φορά μας παίρνει ο χρόνος, παρασυρώμαστε όταν έχουμε πολλά να πούμε. Ε, θα προτιμούσα ε, να τονίσουμε τα θετικά σημεία. Ε, τόνισε και ο συνάδελφος Ρώση ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη δημογραφική αλλαγή Υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία ε, δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση ε, και υπάρχουν στοιχεία τα οποία καλώς δεν συμπεριλαμβάνονται στην ε, έκθεση και η ηλικία δεν είναι ασθένεια. Υπάρχουν πολλά θετικά σημεία τα οποία πρέπει να τονίσουμε και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Όπως είπε και η Γιολάντα Χίμπνερ, τα πανεπιστήμια για την τρίτη ηλικία παραδείγματος χάρη ένα μέτρο θα ήταν η σταδιακή αποχώρηση από την εργασία, ώστε να μπορούν οι ηλικιωμένοι να συνεχίσουν να εργάζονται λιγότερες ώρες. Υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούμε θετικά να αναφέρουμε. γιατί πιστεύω ότι λόγω της ιατρικής προόδου και λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας είναι πολλά τα θετικά σημεία, είναι πολλές οι καινούργιες ιδέες τις οποίες θα μπορούσαμε να προσφέρουμε. Στο 1,5 λεπτό όμως δεν φτάνει, δεν, έχω το χρόνο για να τα πω όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την ηθηγήτρια για την πολύ καλή έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον ε, του, ασθενού, του ηλικιωμένου και ε, ε, χρειαζόμαστε όχι μόνο τεχνικές εξελίξεις αλλά και κοινωνικο-οικονομικές καινοτομίες για να μπορέσουμε να έχουμε ενεργό γύρανση. Στα περισσότερα κράτη-μέλη υπάρχουν διάφορα μοντέλα περίθαλψης ε, τα οποία πολλές φορές ε, είναι παρόμοια ε, και καλό θα ήταν να έχουμε και κάποια νέα στοιχεία, κάποιες καινοτομίες ώστε να μην είναι τυποποιημένες οι λύσεις που προσφέρονται αλλά να υπάρχουν και νέες ιδέες και να δημιουργηθούν και νέα κέντρα τα οποία θα έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Σοφία Κονή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίζω το έργο της εισηγήτριας. Αποτελεί μια εξαίρετη βάση για να δουλέψουμε πάνω. Έχω όμως δύο-τρία στοιχεία που θέλω να αναφέρω και θα υποβάλω και τροπολογία σχετικά. Το πρώτο έχει να κάνει με τον αθλητισμό και την φυσική δραστηριότητα. Στην έκθεση αυτή πουθενά δεν αναφέρεται η φυσική άσκηση η σωματική άσκηση. Πιστεύω ότι είναι κάτι σημαντικό όμως. Λέει η συγγήτρια ότι η ενεργός ε, γύρανση και η υγιής γύρανση προετοιμάζεται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής μας. Ενώ λοιπόν, αν λάβουμε μάλιστα υπόψη μας ότι ο αθλητισμός αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την συνθήκη της Λισαβόνας, ε, πρέπει να το πούμε εδώ, γιατί αποτελεί εργαλείο για καλή υγεία, αλλά αποτελεί επίσης και ένα βοήθημα για κοινωνική επαφή. Έτσι αποφεύγουν την απομόνωση οι ηλικιωμένοι και τη μοναξιά, εφόσον συμμετέχουν σε μια ομάδα που ασκείται σωματικά. Τώρα, δεν είναι το θέμα της ε, οικογενειακής ε, σχέσης. Οι ηλικιωμένοι που είναι σε καλή ε, υγεία, σε καλή κατάσταση, μπορούν να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν τις γενιές οι οποίες είναι ακόμα δραστήριες. Το τρίτο είναι η προσαρμογή των κατοικιών. Γιατί να μην κάνουμε όπως κάναμε για την ενεργειακή απόδοση, να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια για να βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθεί η προσαρμογή των ε, κατοικιών έτσι ώστε να μπορούν αυτόνομα και ανεξάρτητα να ζουν μέσα εκεί οι ηλικιωμένοι. Η Επιτροπή τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την έκθεση. Η Κομισιόν έχει πράγματι προσπαθήσει με αυτή την καινοτόμα πρωτοβουλία να διαφοροποιηθεί από τον πυροματισμό, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή την κοινοτομία όχι μόνο ως τεχνολογική δυνατότητα, αλλά να διερευνηθούν οι δυνατότητες για κοινωνική καινοτομία και έτσι να εξετάσουμε τα συστήματα που πρέπει να τροποποιήσουμε ώστε να απορροφήσουμε την πιθανή ε, αυτή καινοτομία, τεχνολογία ή ιδέες. Έχουμε λοιπόν τριπλό στόχο. Πρώτον, να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη και ζωής και υγείας των πολιτών. Να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των συστημάτων, να είμαστε πιο αλληλέγγυοι επίσης. Και τρίτος στόχος αφορά τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων, νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και για τις αγορές μας, με την έννοια ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης στον τομέα αυτό, που είναι και ένα νέο δυναμικό και, νέα, και για ευκαιρίες. Μπορούμε δηλαδή ε, να έχουμε τριπλά ωφέλη δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε νέα χρήματα, δεν πρόκειται για νέο χρηματοπιστωτικό μέσο. Η ιδέα είναι μέσω τη εταιρική σχέση, είναι ότι κάνοντα πράγματα με νέο τρόπο, προσπαθώντας να βελτιώσουμε την χρήση των υπαρχών των πόρων και να δημιουργήσουμε όσο γίνεται περισσότερες ε, συνεργασίες ώστε να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα. Εμεί λαμβάνουμε Λάβαμε εντυπωσιακό αριθμό απαντήσεων. 261 δεσμεύσεις από διάφορους ομίλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι θέλουν δηλαδή να κάνουν τέτοιου είδους δράσεις. Θέλουν να δεσμευτούν ότι θα κάνουν δράσεις ώστε να αλλάξουν και να δώσουν γρήγορα αποτελέσματα. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το στρατηγικό πλάνο το οποίο φτιάξαμε στην Κομισιόν που εξετάζει συγκεκριμένες δράσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Και οι έξι δράσεις που έχουν εντοπιστεί αφορούν τον τρόπο ε, αγωγής και τον τρόπο συνταγογράφησης. Πολλοί ηλικιωμένοι έχουν πολλαπλές χρόνιες ασθένειες, χρημένοι πολλαπλές αγωγές. Αυτό είναι δαπανηρό ε, και υποφέρουν ταυτόχρονα από παρενέργειες. Το δεύτερο είναι να παρεμποδιστούν οι πτώσεις. Οι πτώσεις ε, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο μετά τα 65 έτη. Δημιουργεί μεγάλο κόστος για τα συστήματα Τρίτος, το άλλο στόχος είναι η αποφυγή της παρακμής της λειτουργικότητας των ανθρώπων. Χρειάζεται να λειτουργούν ακόμα και αν έχουν κάποιο είδος αναπηρίας. Ε, τέταρτη δράση είναι να δημιουργηθεί ολοκληρωμένο σύστημα υγείας και γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο ε, ε, Εξίσου να προωθήσουμε τη δραστήρια και ανεξάρτητη ζωή όχι μόνο για ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες αλλά και για φυσιολογικούς ε, ανθρώπους που πρέπει να χρησιμοποιήσουν το δυναμικό που υπάρχει στην αγορά για να είναι πιο δραστήριοι και να ζουν με, μια καλή ποιότητα ζωής. Ο έκτος στόχος είναι να δημιουργηθεί να δημιουργηθεί περιβάλλον φιλικό προς τους ηλικιωμένους, δηλαδή πόλεις ε, και μέσα μεταφοράς φιλικά προς τους ηλικιωμένους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα φυσικά, ε, μιλάμε για συγκεκριμένες δράσεις, για αυτές τις ε, τομείς δράσης. Τώρα, αναφέρατε και ήδη ρωτήθηκε και η Κομισιόν αν υπάρχουν εμπόδια. Ναι, υπάρχουν πολλά εμπόδια και αυτή η ιδέα της εταιρική σχέσης ε, σημαίνει πως οι εταίροι θα βοηθήσουν για να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά. Ένα από αυτά τα εμπόδια είναι, για παράδειγμα, η έλλειψη διαλειτουργικότητας των συστημάτων μας. Ορισμένες συσκευές μπορούν να δουλέψουν σε μια περιφέρεια μια χώρα, αλλά όχι σε ολόκληρη την Ένωση. Οπότε, ε, μια από τις πρώτες προκλήσεις είναι τα πράγματα να μπορούν να λειτουργούν παντού στην ευρωπαϊκή αγορά. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Ένα είναι το ε, Φλάντρις και που αναφέρθηκε. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα σε περιφερειακό επίπεδο. Η Σκοτία π.χ. είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιείται ολοκληρωμένη βοήθεια για το μεμπομονωμένο πληθυσμό. Έχουν πολύ μεγάλο αριθμό τέτοιου πληθυσμού. Και δεύτερον, να εντοπίζεται ο πληθυσμό που μπορεί να είναι ευαίσθητος σε πτώσεις και να αποφευχθούν οι πτώσεις ή να αποφευχθούν οι άνθρωποι οι οποίοι υποσυτίζονται. Άνθρωποι που στην πλούσια Ευρώπη ζουν και πεθαίνουν στα νοσοκομεία λόγω της, του υποσυτισμού. Και αυτό είναι εύκολο να το αντιμετωπίσουμε αν χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες και την τεχνολογία που έχουμε για να εντοπίζουμε εκ των προτέρων. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα για το τι συμβαίνει ε, Αυτό στο τοπικό και σε περιφερειακά επίπεδα. Σήμερα γίνεται μια μεγάλη διάσκεψη με 450 εταίρους όπου εξηγούν τι κάνουν και τι θέλουν να κάνουν μαζί σε συνεργασία ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί συνδυάζοντας τους πόρους τους. Ευχαριστώ πολύ. Η συγκήτρια μήπως θέλει να λάβει και πάλι το λόγο. Ναι, Θέλω, σύντομα θα αντιδράσω. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ όλους σας που μιλήσατε ε, για την ε, πρόληψη, για τον αθλητισμό, την ε, κίνηση. Ναι, πρέπει, όντως. Άκουσα πάρα πολλές προτάσεις δηλαδή και σας ευχαριστώ ειλικρινά πολύ. Με ενθαρρύνεται έτσι να εμπλουτίσω την έκθεσή μου με τροπολογίες. Έχω μια παρατήρηση να κάνω γιατί διάφοροι συνάδελφοι είπαν ότι πρέπει να τονίσουμε την καινοτομία στην φροντίδα, στην περίθαλψη. Μόνο εκεί. Για μένα όχι. Δεν πρέπει μόνο εκεί να βάλουμε την καινοτομία. Όχι, όπως λέει και η Επιτροπή, πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα φιλικό προς τους ηλικιωμένους περιβάλλον. Η Επιτροπή λοιπόν πρέπει να υπογραμμίσει και το περιβάλλον και την ασφάλεια των τροφίμων, που στο κάτω-κάτω είναι δικές μας αρμοδιότητες. Γι' αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό και να μην το παραβλέψουμε. Ε, και κάτι τώρα για την διαθροτική προσέγγιση των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων. Αυτό έρχεται από τις εργασίες της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Έτσι κι αλλιώς, αυτό που πρέπει να φροντίσουμε είναι να μην φτάνουν στο όριο της στόχιας οι άνθρωποι. Δηλαδή να μην υπάρξει τέτοια μείωση των επιδομάτων, των συντάξεων των ανθρώπων, ώστε τελικά στα γερατιά τους ή και όχι στα γερατιά τους καταλήγουν οι άνθρωποι να παραβλέπουν την υγεία τους γιατί δεν έχουν αρκετά χρήματα. Αυτό πρέπει να το δούμε πολύ και την κοινοτομία να την δούμε και στις πόλεις και στο περιβάλλον και η καινοτομία αυτή μπορεί να βοηθήσει και για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης, οπότε να δώσει οικονομική όθηση και όχι να μας αφήσει σε ένα σπιράλ προς τα κάτω. Σίγουρα με τις παρατηρήσεις σας και με τις σκέψεις σας θα εμπλουτίσω την έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λιωτάρτη. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 23 Νοεμβρίου και μετά στις 18 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε και θα φτάσει στην Ολομέλεια μάλλον τον Φεβρουάριο του 2013. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης θα το αναλάβει η συνάδελφος ε, Κρίστα Κλάς. Θα έρθει στην Προεδρία. Ναι, σε μηδέν λεπτά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το τελευταίο σημείο της μερίσιας διάταξης, αλλά ελπίζω ότι θα με δώσουν λίγο περισσότερο χρόνο οι διερμηνείς. Θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο ε, κύριο Ρεστερόση. Το θέμα είναι η βελτίωση των ωφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης. Σας ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί έχει ήδη τελειώσει ο χρόνος μας. Το θέμα αφορά την αποκόμιδη των καλύτερων δυνατών ωφελών για κάτι το μάλλον από την νομοθεσία που υπάρχει για την ε, κοινοτική νομοθεσία εννοώ, για την προστασία του περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, αν και έχω την αντίρρηση ότι δεν έχει γίνει καμιά αναφορά στις τοπικές αρχές. Ε, να θυμίσω στους συναδέλφους πως συχνά οι σε αυτέ οι τοπικέ αρχέ είναι αυτέ που επιτρέπουν τι ή κάνουν, την εγκατάσταση ή κάνουν του ελέγχου, Γι' αυτό και θα πρέπει να τους έχουμε περίπου. Συχνά δε η εφαρμογή των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων ε, σημαίνουν με σημαντική διοικητική και οικονομική δέσμευση. Γι' αυτό όταν φτιάχνουμε νόμου θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στους περιπαλαιωμένου ε, που πρέπει να καταργηθούν αλλά από την άλλη πλευρά να φτιάχνουμε και ε, απλούς ε, ευνόητους κανόνες εφαρμόσιμους με το λιγότερο δυνατό κόστος υπησβάρος των εταιριών. Ε, σύντομη αναφορά στην, στην δικαιοσύνη την περιβαλλοντική και εδώ εκφράζω τη λύπη μου γιατί η οδηγία η περιπρόσβαση του κοινού στα θέματα δικαιοσύνης για το περιβάλλον είναι αυτή τη στιγμή μπλοκαρισμένη. Ελπίζω πως θα μπορέσει να προχωρήσει γίνεται πιο σύντομα και αυτή η ε, διάταξη. Ευχαριστούμε κύριε Σίτα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σύντομος. Θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο και στους κοιόδης συζητητές. Δεν έχουμε όμως καθόλου χρόνο. Έχουμε και μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 5η Δεκεμβρίου και η κατάθεση τροπολογιών, η κατάθεση τροπολογιών μέχρι Νοεμβρίου και η δεύτερη συζήτηση στις 5 ε, Νοεμβρίου. Ο κύριος Καρλ Φλόρενς. Ε, πρόεδρε, δεν είμαι ικανοποιημένο με την παρουσίαση και με την έκθεση του συναδέλφου Ρώση, γιατί όταν σκέφτεται κανεί τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη για την υλοποίηση των θεμάτων αυτών, τι να πω, θα έγραφε κανείς σελίδες επί σελίδων και θα έπρεπε να γράψει κανείς κάποια κριτική επί των προβλημάτων. Πού βρίσκονται τα προβλήματα. Αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα για τις τοπικές και περιφερειακές ε, ε, κοινότητες. Δεν δώσατε καμιά απάντηση σε αυτό το θέμα, κύριε Ρώση. Λέτε ότι έχουν προβλήματα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποια, πείτε τα. Θέλετε να υπερασπιστείτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίτε μας πού είναι τα προβλήματα, πού πρέπει να αλλάξει κάτι. Στο REACH πρέπει να αλλάξει κάτι. Πού πρέπει να αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι δεν θέσατε το δάκτυλο επί τον των ύλων ήλων και νομίζω ότι ε, και αυτό και με την επικουρικότητα ε, μπορεί να το επαναλάβει κανείς. Λέτε ότι ο σαφής προσδιορισμό κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί προβλήματα. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Και νομίζω ότι και τα θέματα μεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας ακριβώς είναι παράδειγμα για το ότι θα έπρεπε το αντίστροφο να ισχύει από αυτό το οποίο υπενήσεστε. Ευχαριστώ να βοηθήσω ίσως να προσφέρω βοήθεια. Και στο άρθρο 4, αν σωστά καταλαβαίνω αυτό το άρθρο, γιατί στη μετάφρασή του το βλέπω πολύ πολύπλοκο, τι περιμένετε ότι η Ευρώπη θα καταβάλει χρήματα για να τα υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα των σκουπιδιών τα σκουπίδια από το Μιλάνο έρχονται στην περιοχή του Ρουρ, στη Γερμανία. Κάτι θα πρέπει να εφαρμοστεί εφόσον υπάρχει η κοινοτική νομοθεσία. Και αν τυχόν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κοινοτική νομοθεσία, πείτε το και βοηθήστε να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά πριν με χτυπήσει η πρόεδρο με το σφυράκι τη, νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσω εδώ την παρέμβασή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Καρλ Χάιν Φλόρεν. Δεν έχουμε χρόνο, όπω είπαμε. Θα δώσω το λόγο και στο Γιώλα Λάινεν. και η Σάτου χάσει από τους κοιόδης συζητητές. Τζούτι Γκέρλιν και η Σοφία Κονή, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να λάβετε το λόγο στην επόμενη συζήτηση επί του θέματος, ο Γιώργο Λάινεν. Θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι μια σημαντική έκθεση γιατί στυλιτεύεται η ελληπής εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και για το περιβάλλον και για την οικονομία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ε, ε, επενδύσεων που δεν ε, περατώνονται, που δεν φτάνουν στον σκοπό τους. Όπως είπε και ο Καλ Χάινς Φλόρεντ, δεν φταίει το περιβαλλοντικό δίκαιο, φταίει η ελληπής εφαρμογή του στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε διάφορα επίπεδα. Ο Δόκτωρ Στόιμπερ στην Επιτροπή μας είχε πει ότι ο ίδιος νόμος, η ίδια διάταξη, ο ίδιος κανονισμός εφαρμόζεται σε μια χώρα, ενώ σε μια άλλη περιοχή της ίδιας χώρας, σε μια άλλη χώρα, ε, δεν εφαρμόζεται. Χρειαζόμαστε κάποιους μηχανισμούς για να βελτιωθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας. και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο αναφέρει τα ελλείμματα που υπάρχουν. Θα πρέπει να θεσπιστούν όλοι οι μηχανισμοί και όλα τα εργαλεία συγκεκριμένα, οπω είπε ο Καρλ Χάιντς Φλόρενς, για να δούμε πώ μπορούμε στην πράξη ε, να βελτιώσουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σα του χάσει. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτό το έγγραφο εργασίας. Συμφωνώ και με τον Καλ Χάινς Φλόρες και με τον Λάινεν για την ανάγκη βελτίωσης της κατάστασης. Στην έκθεση αυτή ο εισηγητής τονίζει το ρόλο των τοπικών αρχών, την ανεπάρκεια μάλλον του ρόλου των τοπικών αρχών για την αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι προτάσεις της Κομισιόν προχωρούν προς σωστή κατεύθυνση, συμπαριλαμβανομένες της συλλογή στοιχείων με τρόπο που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους στόχους. Χρειάζεται κάποια προσπάθεια ώστε η νομοθεσία αυτή να καταστεί σαφέστερη για τους πολιτές ώστε να μπορούν όντως να ωφεληθούν από την εφαρμογή της. Συγκεκριμένα, στην καθημερινή του ζωή. Συχνά όταν ε, μάλλον αυτή τη στιγμή ρυθμίζεται ένα πρόβλημα, ο κόσμος το ξεχνά πια. Για παράδειγμα, στη χώρα μου, μιλάμε για την νέα νομοθεσία για το ναυσιπλοεία και την ε, όξυνση των, ε, την, ε, τα όξινα ύδατα, την ρήψη θείου. Ε, πριν από κάποια χρόνια είχα διαβάσει σχετικές εκθέσεις ε, για τις λίμνες ε, επίσης. Ευχαριστούμε κυρία Χάση. Ζητώ συγγνώμη από όλους, αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Θα σας δώσουμε περισσότερο χρόνο στην επόμενη συζήτηση. Έχουμε και την Επιτροπή σήμερα μαζί μας. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, όπως είπα, και την Επιτροπή θα ήθελα να παρακαλέσω να αναβάλει την παρέμβασή της μέχρι την επόμενη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι συμφωνείτε. Ελπίζω να συμφωνεί και ο εισηγητής. Να κλείσουμε τώρα τη συζήτηση. Και σας ευχαριστώ όλους. Στις 28 Νοεμβρίου θα γίνει η επόμενη συζήτηση για αυτό το θέμα και θα προτιμήσουμε, θα δώσουμε ε, κατά προτίμηση το λόγο σε αυτούς που σήμερα δεν μπόρεσαν να μιλήσουν. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και τους διερμηνείς που μας έδωσαν περισσότερο χρόνο και θα τα ξαναπούμε στην επόμενη συνεδρίαση στις 12 Νοεμβρίου.